όσον αφορά το υπερσιασμό του δυναμικού ταγουγού Nord Stream και επιπτώσεις στην Ενεργειακή Ένωση και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Δίνω το λόγο εν ονόματι του Συμβουλίου στον Υπουργό, τον κύριο Νικολά Σμιτ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, η όρια ασφάλειας εφοδιασμού στον τομέα της ενέργειας απαιτεί πιο στενή συνεργασία και στο εσωτερικό μα αλλά και με τους εταίρους μας. Κάτι το οποίο βρίσκεται ψηλά ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι είναι και στρατηγική σημασία η ενέργεια και η ασφάλεια εφοδιασμού αποτελεί ένα τεράστιο διακύδευμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, πολλά μέτρα έχουν ήδη ληφθεί από το παρελθόν. Για παράδειγμα, το τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά, η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή αποτελεσματικότητα η οποία ενισχύει την ανεξαρτησία μας και οι προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την συνεργασία με γείτονες της ενέργειας. Το 2014 η Ενεργειακή Ένωση μπήκε στο αυλάκι. Η Προεδρία πιστεύει ότι ήταν πολύ σημαντικό στάδιο, ένα ποιοτικό άλμα στην ανάπτυξη, εκπόνηση μιας νοσιακής ενεργειακής πολιτικής και ασφάλεια εφοδιασμού. Έχει πέντε διαστάσεις πολύ σημαντικές ασφάλεια εφοδιασμού, εσωτερική αγορά ενέργειας, αποτελεσματικότητα στο τομέα της ενέργειας, μείωση των εκπομπών και τέλος έρευνα και καινοτομία. Γι' αυτό το τελευταίο σημείο θέλω να υπενθυμίσω ότι η Προεδρία οργάνωσε στο Λουξεμβούργο πρόσφατα την εβδομάδα της ενεργειακής τεχνολογίας, όπου συγκεντρώθηκαν πάνω από 500 δήμονες του τομέα, Υπουργοί Ενέργειας και επικεφαλής ε, επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρηματίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ενεργειακή Ένωση προωθεί την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας. Συνεργασία η οποία θα επιτρέψει να ενισχύσουμε την ολοκλήρωση των αγορών, προσφέροντας και εξοικονομήσεις αλλά και νέες επενδύσεις. Προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η Ενεργειακή Ένωση, χρειάζεται να ενισχυθεί και η ασφάλεια εφοδιασμού, όπως είπαμε. Γι' αυτό περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016, νομίζω, σύνολο προτάσεων για τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο. Η Προεδρία παρακολουθεί τις προπαρασκευαστικές εργασίες και σε επίπεδο δημόσιας διαβούλευσης για αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα το σχέδιο επέκτασης του δυναμικού του Nord Stream. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα δεν έχει εγκρίνει επίσημα τη θέση της. Πρόκειται για ένα εμπορικό σχέδιο μεταξύ ρωσικών επιχειρήσεων και θετικών επιχειρήσεων. Η Προεδρία αντιλαμβάνεται ότι το σχέδιο αυτό έχει διαστάσεις και ενεργειακές και οικονομικές και πολιτικές και περιβαλλοντικές και ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ε, συνεισφορά στη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, αλλά έχει να κάνει και με τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό σε άλλες χώρες. Κομισιόν που είναι θεματοφύλακα των συνθήκων έχει ως καθήκον να εξετάσει το σχέδιο αυτό στα πλαίσια του νομοθετικού πλαισίου του εφιστάμενου και βάσει και των κανόνων της εσωτερικής αγοράς. Η Προεδρία από την πλευρά της σας διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί το Συμβούλιο την υπόθεση αυτή και συγχρόνως συνεχίζει να προχωράει με την εφαρμογή της Ενεργειακής Ένωσης και την ενίσχυση κυρίως της ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς επίσης και με την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας συγχρόνως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούσαμε σήμερα πολλά μηνύματα για το κλίμα. Οι ανανεώσιμες λοιπόν πηγές ενέργειας έχουν άμεση σχέση με αυτό ακριβώς το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Το λόγο τώρα έχει ο Επίτροπος Μιγέλ Αρία Κανιέτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, επιστρέψτε μου να στείλω ένα μήνυμα και να τον ισχύσω. Πρέπει να έχουμε ασφάλεια, ασφαλή εφοδιασμού για τι πολίτε Ευρωπαϊκή Ενώσεω και για τι εταιρείε. Είναι ύψιστη προτεραιότητα αυτή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στου επόμενου μήνε και μόνο θα προωθήσουμε με θεώρηση τη ασφάλεια του κανονισμού για την ασφαλή εφοδιασμό φυσικό αέριου. Θα έχουμε και στρατηγική για το υγροποιημένο αέριο και αποθήκευση και στι διακυβερνητικέ συμφωνίε θα επιφέρουμε αλλαγέ για να ευθυγραμμίζονται στου στόχου ασφαλού εφοδιασμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και γι' αυτό επίση έχουμε δεσμευτεί να έχουμε επίκυλε μορφέ ε, ενεργείας και διαδρομές και πηγές. Δεν θα πρέπει να εξαρτώμαστε από ένα δρόμο και έναν προμηθευτή. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πολλές πηγές φυσικού αερίου. Είτε είναι από αγωγό, από διαφορετικές πηγές, υγροποιημένο αέριο, υποθηκευμένο αέριο. Λοιπόν, θέλουμε, έχουμε μια αυξανόμενη ενεργειακή αγορά. Θα μας επιτρέψει να μειώσουμε τις ε, να φτάσουμε από 40 εκατομμύρια κυβικά μέτρα στα 90 κυβικά, ε, εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Θα επιταχύνουμε και καλύτερη διασύνδεση μεταξύ κρατών μελών. Έχουμε προχωρήσει αρκετά εκεί. Τους τελευταίους μήνες και μόνο καταφέραμε να έχουμε πρώτα απτά αποτελέσματα στις περιοχές εκείνες που ήταν ανεπαρκώς καλυμμένες και συνδεδεμένες με την εσωτερική αγορά. Να δώσω κάποια παραδείγματα. Η νέα ομάδα υψηλού επίπεδου για τη συνδεσιμότητα ε, στην νοτιοδυτική Ευρώπη για το αέριο θα αυξήσει τι συνέσει ε, στην εποχή μετά το South Stream. Η πολιτική συμφωνία μεταξύ Ισπανία, Πορτογαλία ε, και Γαλλία για τον αρμόδιο αγωγό, θα αυξήσει τη διασύνδεση φυσικό αέριο μεταξύ Βυρική Χερσονήσου και την υπόλοιπη Ευρώπη και ελπίζουμε ότι θα λειτουργεί πλήρω αγωγό μέχρι το 2020. Επίση έχει δομολογηθεί δουλειά για 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο φυσικό αέριο από το Αζερβαϊτζάν στην Ευρώπη το 2020 μέσω τη ανατολική Ογωγού και από αυτή που διέχεται από την Αδριατική. Θα πρέπει να υπάρχει και άλλη διασύνδεση που θα είναι βασικό εργαλείο που θα ολοκληρώσει και τι βαλτικέ χώρε τι εντάξει στην Ευρώπη. Την επόμενη εβδομάδα θα φροντίσουμε τελικά να καρποφορήσει αυτό. Θα έχουμε τη συμφωνία για τον διασύνδεση GIPL μεταξύ Πολωνία και Λιθουανία και θα υπογραφεί σχετική συμφωνία. Οπότε θα συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και περίπου στο ύψο των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν μπορώ να τον παρανατονίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό, διότι ω έχουν τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα ε, εξαρτάται από, το αέριο της Ρωσίας και περίπου το μισό από αυτό περνά από την Ουκρανία. Και εδώ έρχομαι στο Nord Stream 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε δεόντως ε, τη συμφωνία των μετόχων να ε, επεκταθεί ο αγωγός Nord Stream το πρώτο που θα πούμε είναι το Nord Stream 2 παραμένει ένα εμπορικό πρόγραμμα και βεβαίως εμείς είμαστε εμπορικό μέρος και θα κατασκευάσουμε τις υποδομές. Αλλά πρέπει να τονίσω όπως οποιοδήποτε άλλο αγωγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτός ο αγωγός θα πρέπει να σέβεται απολύτως τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεω και κυρίως το τρίτο ενεργειακό πακέτο καθώς και θέματα περιβαλλοντικά θέματα ανταγωνισμού και δημοσίων προμηθειών, κατοικών προμηθειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, αυστηρά θα προβεί στην αξιολόγηση, θα συγκρίνει κατά πόσο συμμορφώνεται με το, θεσμι... με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Και θα γίνεται λοιπόν η σωστή αξιολόγηση. Η δυνατότητα μεταφορών από τη Ρωσία ε, χρησιμοποιείται μόνο κατά 50% και αυτό ήδη ξεπερνά τι ανάγκε Ευρωπαϊκή Ενώσεω για μελλοντικό φοδιασμό. Αν κατασκευαστεί το Nord Stream 2, σύμφωνα με τι εκτιμήσει μα, θα αυξήσει τι δυνατότητε διαβίβαση από τη Ρωσία θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργά υποστηρίζει τι προσπάθειε ούτω ώστε εξασφαλίζεται ότι η Ουκρανία είναι και θα παραμείνει σταθερό και αξιόπιστος, ε, αξιόπιστη χώρα διέλευση. Να υπογραμμίσω εκ νέου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανοιχτή για το ρωσικό αέριο και θα ήθελε η Ρωσία να είναι ένα αξιόπιστο προμηθευτή φυσικού αερίου στο μέλλον. Αλλά επίση και η μεταφορά του ρωσικού αερίου θα πρέπει να μπορεί να ταιριάξει στη δική μα τη ποικιλομορφία. Και ότι ο ρωσικό προμηθευτή, όπω άλλο προμηθευτή Ευρωπαϊκή Ενώσεω, θα, θα συμμορφώνεται με του κανόνε περί ε, αγορά, εσωτερικής και ανταγωνισμού. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ξεκινάμε τη συζήτηση με παρεμβάσεις των εκπροσώπων των ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο Πρόεδρος Μπούζεκ έχει το λόγο. Να σε ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Σέβομαι την ελευθερία του επιχειρήν στα οικονομικά θέματα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να σημειώνουν κέρδη και πρέπει να είναι σεβαστό το νομικό πλαίσιο. Στο Nord Stream 2 έχουμε αμφιβολίες και για την πρώτη συνιστόσα και για τη δεύτερη. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς λόγο για κέρδη, διότι οι ήδη υφιστάμενες υποδομές μόνο κατά το ίμιση χρησιμοποιούνται και αγωγή υπό τον πυθμένα της ε, θάλασσας είναι πολύ δαπανηρότερη από ό,τι αγωγή μέσω ε, της ε, ξηράς, μέσω χερσαίων εδαφών. Και δεύτερον, δεν συνάδουν όλα αυτά με τις υποχρεώσεις ε, για την οικολογική ασφάλεια. Υποχρεώσεις δηλαδή των κρατών μελών να σέβονται το περιβάλλον και την οικολογική ασφάλεια. Και ένας θα έχει το πάνω χέρι. Και υπάρχει εδώ μια διακρύβωση για αντιμονοπολιακές δράσεις κατά της ε, Gazprom από τις ε, ευρωπαϊκές αρχές. Συνοψίζω, αυτό το εγχείρημα δεν μπορεί να θεωρείται καθαρά εμπορικού χαρακτήρα εγχείρημα διότι οδηγεί σε πολιτική, πολιτικές εντάσεις ε, που πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υφίστανται και είναι, αποτελεί κίνδυνο και για τους εταίρους μας ε, στην ε, πολιτική γειτονία στις όμορες χώρες. Ε, αυτό το εγχείρημα μας διχάζει, δεν μας συνενώνει και οικονομικά δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί ποιο είναι το όφελος. Αναμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει όλα τα βήματα και διαβήματα σε περίπτωση μη υλοποίηση των όρων και προϋποθέσεων από πλευράς ε, του North 2 και να υπάρξουν και οι συνέπειες ακριβώς όπως και με το North Stream 1. Ευχαριστώ. Κύριε Μπούζεκ, υπάρχει μια ερώτηση για σας. Θέλετε να την ε, απαντήσετε. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει το λόγο κύριε Μπάλτσο. Μπάλτσο. μικρόφωνο. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, ο North Stream πρόκειται να παράσχει ρωσικό αέριο στη Γερμανία άμεσα και είπατε ότι σήμερα δεν εξοπλίζει όλε οι δυνατότητε. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε επομένως έναν καινούριο αγωγό. Οπότε και έτσι θα έχουμε διπλασιασμό της παροχής. Δεν συμφωνείτε ότι με αυτή την παραπάνω παροχή πρόκειται η Γερμανία να είναι σε ετοιμότητα για το μέλλον όταν δεν θα παίρνει φυσικό αέριο από την Ουκρανία. Μπα και αυτό προετοιμάζει η Γερμανία. Μπούζεκ. Και εδώ πρέπει να πω σε σχέση... ...są wykorzystywane tylko εδώ σε σχέση με τη διασύνδεση μόνο κατά 50% υπάρχει εδώ αύξηση σε σχέση με το δυναμικό, το υφιστάμενο δυναμικό των ε, ενισχύ διασυνδέσεων. Γι' αυτό αυτή η ε, δημιουργία, αυτό το εγχείρημα είναι απόλυτα περιττή μια και η ήδη υφιστάμενη διασύνδεση δεν αποτελεί στο 100% αντικείμενο εκμετάλλευσης ακόμα. Νάτο. In nome del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici. Ο κύριο Τζανονάτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε, μα ανησυχεί και μα ανησυχεί πολύ το ότι τώρα θα διπλασιαστεί η δυνατότητα παροχή του Nord Stream. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, ακριβώ όπω ελέγχθη, πρόκειται να αυξήσουμε την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Και έτσι ε, θα, θα υπάρξει ε, διέλευση από αυτές τις τρεις χώρες ε, για το Nord Stream. Τώρα θα υπάρχει διπλάσια παροχή επομένω. Οπότε θα έχουμε και διέλευση του αγωγού και από τη Λευκορωσία και από την Ουκρανία, εκτός από τη Ρωσία. Οπότε έτσι δεν θα έχουμε κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά την παροχή. Οπότε ήδη θα είναι ακόμα χειρότερη η αρνητική ισορροπία δυνάμεων σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε θα πρέπει έτσι να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιο είδους πιο φιλόδοξη διακυβέρνηση όσον αφορά την πολιτική ενέργειας. Γιατί η, ασφάλεια της παροχής είναι κάτι πολύ βασικό. Και είναι, επομένως θα πρέπει να δούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνει όσον αφορά αυτή την ενεργειακή πολιτική. Γιατί ε, έτσι τώρα εάν έχουμε την Ουκρανία σε αυτή τη διαδρομή σημαίνει ότι αυτή η χώρα δεν θα μπορέσει να σταθεροποιηθεί και έτσι η χώρα θα είναι υπό την, ε, ε, υπό, υπό την ρωσική εξουσία και έτσι το 2020 θα ολοκληρώσουμε αυτή την διαδρομή και θα έχουμε πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ που θα χαθούν τα οποία τώρα αφορούν αυτούς τους δασμούς διέλευσης. Αυτό είναι απειλή η οικονομική και κοινωνική για τη χώρα εκείνη αλλά επίσης και για την ε, ενέργεια ε, της Ανατολικής Ευρώπης. Εν κατακλείδη πρέπει να σας πω ότι ο South Stream ουσιαστικά από την παρούσα κατάσταση έχει γκρεμιστεί γιατί ακριβώ έχουμε όλες αυτές τις κριτικές ε, που αφορούν τον North Stream για το, την ECR τον, ρόλο, ε, τον λόγο έχει ο κύριος Γκρόμπαρτσικ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγα χρόνια θυμάμαι τον Επίτροπο κύριο Ότιγκερ που έλεγε γιατί οι Γερμανοί συμμετέχουν στην κατασκευή του Nord Stream το κοινοβούλιο ήταν κατά και έλεγε τότε ο Επίτροπος ότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται δεν θα προβούν ξανά σε τέτοια επένδυση και γι' αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω γιατί κύριε Ότιγκερ κάνανε αυτή την κίνηση οι Γερμανοί γιατί θέλουν να κατασκευαστεί αυτή η καινούργια διαδρομή και όταν τον ρώτησα τον ίδιο μου είπε ότι είναι ιδιωτική γερμανική πρωτοβουλία αυτός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γι' αυτό και πριν από λίγες εβδομάδες σας ξαναρώτησα κύριε Επίτροπε τι γίνεται με το North Stream στα πλαίσια του τρίτου ενεργειακού πακέτου της ε, Ένωσης. Έχω αναλάβει και εγώ μια έκθεση σχετικά και εσείς με παραπέμψατε στην απάντηση Έτιγκερ. Είπατε ότι πρόκειται για ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν έχει ουδεμία αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 110 δις κυβικά μέτρα θα δίνει. Δηλαδή 50% ε, της πρώτης ύλης των εισαγωμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως αυτό αντιβαίνει στην ε, πρόταση ε, της διαφοροποίησης της ε, προμήθειας ενέργειας. Μιλούμε για όλες τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης οι οποίες τώρα θα είναι εις το έλεος της προμήθειας ενέργειας από την Ρωσία. Άρα θα πρέπει τα κρατη να αναθεωρήσουν θα πρέπει να αναθεωρηθεί η ενεργειακή πολιτική. Πρόκειται για μια παθητική στάση. Εάν προχωρήσουν οι Γερμανοί σε αυτήν την επένδυση, η διαίρεση και ο διχασμός της Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να γίνει πιο βαθιά. Είναι εδώ να, εκτραπεί έτσι η ενεργειακή μας πολιτική. Για την άλλη. Ο κύριος Πέτερσεν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το έργο North Stream 2 είναι ζωτική σημασία για την ε, ενεργειακή αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για το τρίτο ενεργειακό πακέτο και για την Ενεργειακή Ένωση. Η Ρωσία θα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός εταίρος Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλά χρόνια. Είμαστε, ε, υπάρχει αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε εμά και στη Ρωσία και αυτό φαίνεται και στα έργα που έχουμε κοινά. Η Ρωσία είναι ένας κύριος εξαγωγός φυσικού αερίου και η Gazprom έχει αντιταχθεί στις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς και μάλιστα προσπάθησε να υπονομεύσει ε, αυτήν με τις διάφορες στρατηγικές που ακολούθησε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κάθε λόγο να εφαρμόσουμε ε, το μεγαλύτερο επίπεδο ελέγχου στις ε, πρακτικές τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται πάνω στους στόχους για την ε, μελλοντική ενεργειακή ένωση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα εγώ να μου πείτε τις εκτιμήσεις σας για το πώς θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις συζητήσεις για τον αγωγό North Stream 2 στα πλαίσια μάλιστα των κατευθυντήριων γραμμών. Για παράδειγμα, μπορείτε να μας πείτε πόσα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διεξάγουν στρατηγικές ε, μελέτες που θα εκτιμήσουν τις γεωπολιτικές επιπτώσεις του έργου αυτού. Πιστεύω πως οι περισσότερες χώρες διεξάγουν εκτιμήσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου, εκείνες όμως δεν συμπεριλαμβάνουν και τις ευρύτερες πολιτικές επιπτώσεις αυτού του έργου υποδομής. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισέλθει σε διάλογο με τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη και να υποβάλει αναφορά στο Κοινοβούλιο για το ε, πόσα από αυτά τα κράτη-μέλη θα διεξάγουν γεωπολιτικές εκτιμήσεις αντικτύπου των υποδομών αυτών. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω πώς προσεγγίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές ε, τις, ε, αυτά τα θέματα και τι ε, συμβαίνει αν υπάρχει κάποια γεωπολιτική μελέτη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα σε σχέση με την ε, πολιτική γειτονία και με την Ουκρανία. Για την ΓΚΟΕ, το λόγο έχει ο κύριος Ηλικιώτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο διπλασιασμό του δυναμικού του Βόρειου Αυγού έρχεται ω απάντηση στην αδυναμία τη Ένωση να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τις ελλείψεις που αφορούν την ενεργειακή της ασφάλεια. Εν τούτη, τα κυριότερα προβλήματα που αφορούν τον ενεργειακό ανεφοδιασμό υπάρχουν στον νότο τη Ευρώπη και όχι στο βορρά. Σήμερα πολλοί εκφράζουν ανησυχίε για την ενδυνάμωση του Βορειού αυγού. Αυτό όμω που πρέπει να πραγματικά να ανησυχήσει την Ένωση είναι γιατί ακόμα υπάρχουν μέλη που είναι απομονωμένα στον νότο υπάρχουν μέλη στον νότο κράτη μέλη τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα στην ενεργειακή επάρκεια. Αυτό που πρέπει να προβληματίσει επίση είναι ότι με αυτέ τι εξελίξει περιθωριοποιείται ο νότιο αγωγό και η, Ευρω... η... η Κομισιόν πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο τι εγχώριε ε, ενεργειακέ πηγέ συνεχίζει να παραβλέπει τον ρόλο των κοιτασμάτων που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στην κύπρο αλλά και τα κοιτάσματα που υπάρχουν στην ανατολική μεσόγειο και ευρύτερα στην περιοχή της μεσογείου και της βόρειου αφρικής. αναμένουμε από την ένωση να στηρίξει ενεργειακέ επιδίσεις στην ανατολική μεσόγειο να προωθήσει τη δημιουργία ενός μεσογειακού κόμβου φυσικού αερίου με αγωγούς αλλά και την ανάπτυξη παραγωγής lng παράλληλα ζητάμε να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και να διασφαλίσει προσιτέ τιμέ για του καταναλωτέ. αν γίνουν αυτά κανεί δεν χρειάζεται να ανησυχεί για την ανάπτυξη του βόρειου Αγού. Λοιπόν, ο κύριος Τούρμες έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουτχόφερ, ο οποίος ε, είχε αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ο διπλασιασμός του αγωγού μέχρι τη Γερμανία είναι πολύ κακή ιδέα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το θεωρήσουμε σαν πρόκληση μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ε, γειτονίας. Η πολιτική της ε, Ρωσίας είναι σαφή ε, η Ρωσία θέλει να αποκόψει την Ουκρανία από χώρα διαμετακόμισης και βλέπουμε ότι οι παραδόσεις φυσικού αερίου θα γίνουν πιο δύσκολες και δυστυχώς ε, θα, δεν θα μπορέσουμε παρά να υποσκάψουμε τον ανταγωνισμό. Αυτό τάσεται και κατά των γεωπολιτικών μας συμφερόντων στην Ουκρανία. Είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία του σώματος συμμερίζεται αυτά τα επιχειρήματα. Όμως ε, υπάρχουν πολλά λόμπι. Ε, η, Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εγγενή συμφέροντα και προωθούν τις ομάδες πίεσης μέσα στα πλαίσια των εμπορικών του σχεδίων. Και φυσικά έχουν και τον Φρανσουά Ολάν, την Άγγελα Μέρκελ και τον Ντέιβιτ Κάμερον. Άρα πού βρίσκεται η συνοχή σας στην πολιτική της Ουκρανίας, πού βρίσκεται η αλληλεγγύη σας με τις γείτονες χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Δεν είναι εμπορικό σχέδιο. Είναι πολιτικό και εκρηκτικό, καθώς και διχαστικό σχέδιο. Γι' αυτό θα ήθελα η Επιτροπή να είναι στεναρή και έχουμε το σωστό άνθρωπο εδώ ενώπιόν μας. Θα ήθελα και ο πρόεδρος Τούσκ να ανοίξει ένα νέο δρόμο, Εάν αυτό το πρόγραμμα, το project δεν θα φτάσει στην ατζέντα των επόμενων Συμβουλίων Υπουργών, τότε θα ξεχάσουμε την Ενεργειακή Ένωση της Ευρώπης. Θα ήθελα ο κύριος Κάμερον, η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Ολάντ να μας εξηγήσουν γιατί τάσσονται υπέρ αυτού του ναι. προγράμματος το οποίο θα πρέπει να σταματήσει. για την Ευρώπη της, ε, της άμεσης δημοκρατίας, ο κύριος ε, Ταμπουράνο. Το Nord Stream 2 αποτελεί πραγματικό πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επιληθεί γενικότερα. Προσπαθούμε να φτάσουμε σε μία μετάβαση και γι' αυτό δυστυχώς το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί μία γεωπολιτική λύση μέσα στα πλαίσια μίας επισφαλούς ε, ισορροπίας. Κανένας δεν θα είχε υποστηρίξει το North Stream εάν ήταν άλλες οι εξελίξεις στην Ουκρανία με το νέο ψυχρό πόλεμο και στα δικά μας σύνορα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μία Ευρώπη δημοκρατική και ενωμένη δεν θα πρέπει να προωθήσουμε τα συμφέροντα των ε, μεγάλων πολιεθνικών που δεν τάσσονται υπέρ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις επιχειρήσεις του Νότου. Η κατάσταση αυτή είναι πιο δύσκολη, συνάδελφοι. Τι να πούμε για τις κυρώσεις προς την Ρωσία τι θα πούμε για τις ζημίες που πλήττουν την Ελλάδα και την Ιταλία. Τι θα γίνει με τα κέρδη από το North Stream και τον Ουκρανικό λαό τον ξεχάσαμε. Ας, προσπαθήσαμε, ας προσπαθήσουμε ως σωστοί γιατροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασθενεί να βρούμε λύση. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία Ενεργειακή Ένωση για την απομάκρυνση από τη χρήση του άνθρακα μέσα στα πλαίσια της ε, κλιματικής ασφάλειας, αλλά και μία εξωτερική πολιτική προς την ειρήνη και την καλή γειτονία με όλες τις όμορες χώρες, χωρίς να μας επιβάλλει τι θα κάνουμε κανείς. Πιστεύω ότι ε, ε, όλα τα κράτη-μέλη είναι πριν interpares και έτσι θα πρέπει να θεωρηθούν για την Ευρώπη και για την, ε, των Εθνών και την Ελευθερία, ο κύριος Μπαΐ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να προσέξουμε να μην παρασυρώμαστε γιατί βλέπετε ότι εσείς τελικά τι κάνετε, το, το, το χέρι το οποίο σας αστρέφει να, και αυτό γίνεται και με την Ρωσία, εξάρτηση. Ε, γι' αυτό όλοι μαζί το διαπιστώνουμε ποτέ. Επιτρέψτε μου να σας πω τελικά τι είχε πει ο Ζωμφεργέ, ο πρόεδρος ε, του φορέα για το, για το φυσικό αέριο αλλά και του διεθνούς φορέα. Τα είπε αυτό ο Φιγαρό και τα είχαμε πει την επόμενη μέρα που κλείστηκε η συμφωνία με το South Stream. Αλλά ε, είπε επιλέξει ότι δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να αποσυνθεί από το ρωσικό αέριο και αυτό είναι ε, κάτι το οποίο το ομολόγησε και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού για την Ενέργεια. Θα πρέπει να γνωρίσουμε όμως ότι τελικά η Ουκρανία, η ηγεσία τους που είναι αυτοί οι οποίοι τώρα ε, δεν σταματάνε να κατηγορούν την Ρωσία παρά το ότι εσείς τους ενθαρρύνατε και τελικά δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια αυτού του αγωγού που διασχίζει αυτή τη μεγάλη χώρα που έχει δυνατότητες και η Gazprom πολλές φορές έχει απειλήσει να κλείσει τις βάνες γιατί η, ναι, <clears throat> η νευτογκάζ δεν μπορεί να πληρώσει τα ε, και ε, τις οφείλει τα χρέη της. Και μετά από διμερείς τευνές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, στις 25 να του είπε η Κομισιόν ότι θα δώσει 100 εκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία, ούτως ώστε η Ουκρανία να μπορέσει ε, να έχει ρωσικό αέριο φέτος τον χειμώνα. 100 εκατομμύρια ε, δολάρια. Ε, περιμένετε δολάρια, προτιμάτε δολάρια από τα ευρώ και έτσι θα μπορούσαν να ζεσταθούν οι Ουκρανοί. Ε, όμως ακόμη δεν έχουν μπορέσει να πάρουν τύχη στα χέρια τους γιατί έχουν όλα αυτά τα φρένα στην προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί βλέπουμε ότι ο μεγάλος ιστορικός αδελφός δηλητηριάζεται με αυτό το μίσος. Άρα θα, έτσι είδαμε τι έγινε με όλες τις χώρες Τη Νοτιοανατολικής Ασία και από το South την έχουν αφαιρθεί Βουλγαρία, Σερβία, Ουγγαρία αλλά και Ιταλία και Ελλάδα. Οπότε ε, έχουμε την ε, ENG, τους Γάλλους, έχουμε διάφορες εταιρείε οι οποίε στις 4 ε, Ενάτου υπέγραψαν και το συμβόλαιο τόσο ώστε να φτιάξουν το North Stream υπαριθμών 2. Η Gazprom θα έχει το 51% και 10% θα έχει καθ' μία τις εταιρείε και η γαλλική εταιρεία 9%. Ε, Επί ευκαιρία του Οικονομικού Φόρου του Βλαδιβοστόκ, έτσι θα μπορούμε τώρα να έχουμε την ε, διπλάσια παροχέτευση αερίου. Αλλά εσείς αναγκάσατε την ε, Ρωσία να παραιτηθεί από το South Stream. Τώρα έγινε αυτό το μακρόπνο συμβόλαιο, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να υπάρξει κάποια σταθερότητα στην Ευρώπη αντί για αυτόν τον ψυχρό πόλεμο τον οποίο εσείς ξεκινήσατε. Ο Πρόεδρος. Κύριε Μπαϊ, υπάρχει μια περώτηση για εσάς, θέλετε να απαντήσετε, ναι, λέει. Έχει το λόγο κύριε. Αγαπητέ συνάδελφοι, άκουσα όλους τους επένους για την κασπρόμη σαν τον πιο αξιόπιστο πάροχο στην Ευρώπη. Ναι, θα μπορούσε κανείς να το συλλάβει αυτό, αλλά εσείς πώς εξηγείτε το τι είναι στην Κασπρόμ, ότι είναι η πιο διεφθαρμένη μεγάλη εταιρεία στην Ευρώπη. Βλέπουμε όλα αυτά τα τεράστια κτίρια που ανήκουν ε, σε αυτούς που έχουν τα ενία της εταιρεία, έχουμε αυτές τις σκοτεινές συμφωνίες που κλείνουν και πώς ε, εξηγείται το ότι χρεώνει στην Ουκρανία περισσότερο από όσο χρεώνει στη Γερμανία η Γκασπρόμ, Μπά και αυτό έχει ελαττήρια πολιτικά. Δεν είναι σίγουρα οικονομικό το θέμα. Η τιμή για την Ουκρανία παρά για την ε, Γερμανία. Ε, αν είστε οικονομολόγος και διαμορφώνετε την κρίση σας έτσι, αυτές συνάδελφα, ε, είναι ενδεικτικό αυτό το οποίο λέτε για αυτή σας την εχθρική στάση κατά της Ρωσίας που τόσο συχνά ακούγεται εδώ στο Κοινοβούλιο. Γιατί μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο η Γκασπρόμ ουδέποτε έχει αποτύχει να παράσχει αέριο και όσον αφορά τα διαφορετικά τιμολόγια εξηγείται από το ότι είναι σε υπερεμέρεια τόσο συχνά η Ουκρανία έναντι της Ρωσία. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ποσά τα οποία οφείλονται από την Ουκρανία προς τη Ρωσία. Ο Πρόεδρος Κόρβιν Μίκε. Μίκε γραμμένος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Mm. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο ότι αυτές ε, είναι ιδιωτικές εταιρείες. Και ως ιδιωτικές εταιρείες δραστηριοποιούνται και στη Γερμανία και στην ε, Ρωσία. Ο κύριος Άριας Κανιέτε μας είπε ότι ο δεύτερος αγωγός θα οδηγήσει σε μια διαφοροποίηση της προσφοράς. Ε, σας παρακαλώ, μην γίνεστε γελίος. Κύριε Μπούζακ, Πιστεύω πως ε, εδώ πρόκειται περί τον δεύτερο αγωγό, ο οποίος ενδεχομένως θα μπορέσει να αλλάξει τα δεδομένα στην μεταφορά ενέργειας ε, μέσω της Ουκρανίας. Και εδώ πιστεύω πως πρέπει να σκεφτούμε τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αλλού. Υπάρχουν κέρδη από τις ε, μετοχές, από την ε, Gazprom και γι' αυτό δεν ακούμε πολλά αρνητικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει κάτι. Εσείς όμως έχετε υποχρέωση να προστατεύετε όχι μόνο τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά και τα συμφέροντα των ε, κρατών μελών. Μας είπατε ότι δεν ε, συνιστάτε κάποια απειλή από τον ε, North Stream 2, όμως σας παρακαλώ να μην γίνετε κι εσείς ένας υπεργολάβος της Gazprom. Ο κύριος Κάριντς έχει το λόγο. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μεγάλη αδυναμία στρατηγικά. Εξαρτώμαστε από τις εισαγωγές. Εισαγωγές ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και εξαρτώμαστε από όλους τους παρόχους, κυρίως από τη Ρωσία. Και εδώ είναι το αδύνατο σημείο μας. Όμως υπάρχουν λύσεις και αυτοί, αυτές οι λύσεις είναι να ξαναχτίσουμε την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Έχουμε καταρχάς ως καθήκον να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό, να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να γίνει αυτή η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών. Όμως ο αγωγός North Stream 2 έχει καταφέρει το αντίθετο. Δεν εξυπηρετεί τους ε, τρεις αυτούς ε, σκοπούς ε, Τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυξάνει την εξάρτησή μα από την Ρωσία, μειώνοντα ε, ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό. Έτσι δεν σημειώνεται καμία διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και οδηγείται στο να είναι η Ρωσία ο μοναδικό πάροχο ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ θα είναι οι συνέπειε του διπλασιασμού τη χωρητικότητα του North Stream. Επίση, μέσω αυτή τη πράξη θα απομονωθεί τελείω η Ουκρανία και εμεί, ω Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε καθήκον να στηρίξουμε την Ουκρανία Πρέπει να σταματήσουμε αυτό το έργο. Δεν διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να γίνει πολιτικά. Και η λύση ε, σε αυτό θα ήταν ο αγωγός South Stream, ο οποίος σταμάτησε από πολιτική πρωτοβουλία. Επίσης, μπορούμε νομικά να κινηθούμε, να εξετάσουμε το θέμα, να εξετάσουμε τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους παρόχους τρίτων χωρών, δηλαδή την Gazprom. Gazprom. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπαρτσιούτης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργειακά από την Ρωσία ήταν και ένας από τους κύριους λόγους που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την ενεργειακή Ένωση. Γι' αυτό και γίνονται αυτές οι συμφωνίες. Ο διπλασιασμός της φορτικότητας του North Stream αντιβαίνει στην πολιτική μας της Ενεργειακής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση προσπερνώνται κάποια κράτη-μέλη και απομονώνονται από το υπόλοιπο ευρωπαϊκό δίκτυο παροχής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τι θα απογίνουν αυτά τα κράτη. Ο, χώρες όπως η Λιθουανία, η οποία κατάφερε να δημιουργήσει τον τερματικό σταθμό LG χωρίς βοήθεια οικονομική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα γίνουν οι χώρες αυτές όταν υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν αποφάσεις που ζημιώνουν τις χώρες μας. Οι προσπάθειες που κάνουμε να αυξήσουμε την ενεργειακή μας ανεξαρτησία έρχονται σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι σκανδαλώδες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα δεν έχει λάβει όλες τις πληροφορίες για αυτές τις συμφωνίες προτού αυτές υπογραφούν. Είναι σκάνδαλο, επαναλαμβάνω, και αυτό εγείρει ερωτήματα για την αποδοτικότητα των θεσμών μας. Ο κύριος, ο Φωτίγκα έχει το λόγο. Η κυρία, με συγχωρείτε. Νομίζω ότι το Nord Stream ήταν ένα μέσο πίεσης για τις χώρες ε, στην οποία, στις οποίες ανήκω και εγώ ως προς τη στάση της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας. Βλέπουμε ότι και το Turk Stream θα περιοριστεί και ε, βλέπουμε ότι η προπαγάνδα είχε σοβαρό αντίκτυπο, η ρωσική προπαγάνδα εννοώ. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την προπαγάνδα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τον Ιούλιο πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγραψαν στην Επιτροπή ε, μιλώντας για τον δυνατότητα διπλασιασμού της χωρητικότητας του North Stream. Κύριε Επίτροπε, ε, με εξέπληξε η γραπτή σας απάντηση Εάν αυξήσουμε την χωρητικότητα του φυσικού αγωγού, θα είχαμε να κάνουμε με μία εμπορικού χαρακτήρα απόφαση. Δηλαδή μιλάμε για business as usual. Άρα, με βάση τη γνωμοδότηση πολλών συναδέλφων, θα ήθελα να σας ερωτήσω τα εξής. Με βάση την γεωπολιτική στρατηγική σημασία της Ρωσίας θεωρείται ότι πρόκειται για εμπορικό σχέδιο τη στιγμή που παρακάμπτουμε την Ουκρανία. Δεν θεωρείται ότι το Nord Stream αντιβαίνει στην Ενεργειακή Ένωση της Ευρώπης και την Ενεργειακή Στρατηγική της Ευρώπης. Και τρίτον, Πώς αυτά συμβαδίζουν, δηλαδή ο διπλασιασμός της χωρητικότητας του North Stream και της μείωσης της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία. Σας ευχαριστώ εκ των προτέλων για τις απαντήσεις σας. Ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ανάπτυξη της Ευρώπης της ενέργειας σημαίνει ότι αυτός ο ζωτικής σημασίας ε, στρατηγικός τομέας θα υποταχθεί στους μεγάλους οικονομικούς κολοσσούς από πλευράς υποδομής και από πλευράς της ε, φιλόδοξης ολοκλήρωσης των αγορών. Έχουμε να κάνουμε με το θέμα του ενεργειακού ε, εξοπλισμού εφοδιασμού, με συγχωρείτε. Μιλάμε για την ενεργειακή απομόνωση μένων κρατών μελών. Όλα αυτά θα τα αφήσετε σε δεύτερο πλάνο. Πρόκειται για θέματα που άπτονται της δημοκρατικής ανάλυσης του τομέα της ενέργειας. Η ενέργεια είναι ένα δημόσιο αγαθό. Θα πρέπει να υπεξαιρεθεί από τα μεγάλα μονοπόλια τα οποία αφορά μέσα αυτή η ένωση στον τομέα της ενέργειας. Ο κύριος Τάραντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρωτοβουλία του κ. Σεύτσογλου, ώστε να διερευνήσει τι γίνεται με την νομική πλευρά του Nord Stream 2, είναι κάτι το οποίο το χαιρετίζουμε γιατί νομίζω ότι έτσι ε, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε, ώστε να έχουμε κέρδο στα γεωπολιτικά και επίσης και αυτό είναι ε, κομμάτι από αυτόν τον υβριδικό πόλεμο γιατί όσο και να έχουμε ε, την ευγενή στάση των Ρώσων δικηγόρων της Dutch Shell κλπ. Τελικά, κύριε Κανιέτα, είχατε όλη την πολιτική υποστήριξη για να μπορέσετε να τους υπερκεράσετε και να τους παρακάμψετε όλα αυτά, για να μην βγούμε όλοι χαμένοι, λούς-λούς. Ξέρουμε ότι, ότι τα τρία θεσμικά όργανα ε, και αυτό το, το, τρίγωνο θα γίνει τρίγωνο των, βερμίδων, των, των βερμούδων από θεσμικό τρίγωνο. Οπότε θα πρέπει ο κύριος Τούσκ να αναλάβει δράση. Συγγνώμη, δεν πρόφερα καλά το όνομα του. Ο κύριο Τούσκ να αναλάβει δράση και να μπορέσει το θέμα αυτό να το εντάξει στο θεματολόγιο του Συμβουλίου. Γιατί μόνο τότε η Φράου Μέλκελ και ο Μεσχέ Λόντ θα μπορέσουν να δούνε μέσα από τα μάτια το Σομπότκα, του, όλων αυτών των ε, μαρτύρων, το τι τραγικό λάθος είναι τον κύριο Πούτιν και τον κύριο Σρέντερ να τους βάλουν στο παιχνίδι, να φτιάξουν αυτόν τον αγωγό που δεν είναι βιώσιμος και να καταστρέψουν το περιβάλλον. Κύριε Κανιέτε, εσείς νομίζω ότι έχετε ε, ε, ασχοληθεί με το πετρέλαιο και εγώ με το φυσικό αέριο, γιατί είχα ασχοληθεί στον ε, Σοβιετικό στρατό με αυτές τις, ε, αυτούς τους αγούς που είχαν να κάνουν και με τον Γερμανικό στρατό τελικά. Αυτό είναι μια μεγάλη μπλόφα της Ρωσίας. Και ας έχει κάποια εκατομμύρια να δώσει για τη βιτρίνα στη Γαλλία, αλλά τελικά το 50% πάνε στο Nord Stream 1. Οπότε θα πρέπει να σταματήσει αυτό το, το ηλίθιο πρόγραμμα το οποίο πρόκειται πρώτα απ' όλα να σκοτώσει την Ουκρανία και μετά του υπόλοιπους Μιλήσατε με το διπλάσιο χρόνο από όσο είχατε στη διάθεσή σα, κύριε, λέει ο πρόεδρο. Στον κύριο Τάραντ. Και τώρα, ο κύριο Σένφελτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκυται στο να έχουμε λιγότερη εξάρτηση από την Ανατολική Ευρώπη. Επομένως, δύσκολα κανείς να θεωρήσει ότι αυτός και ο αγωγός ε, συνάδει με τα ενεργειακά μας συμφέροντα και την ενεργειακή μας στρατηγική. Άρα η κατάσταση τώρα είναι αρκετά παράδοξη. Έχουμε αυτά τα στρατηγικά έγγραφα της Ένωσης που τονίζουν το ότι θα πρέπει να υπάρχει πολλαπλότητα, πλουραλισμός όσον αφορά τις πηγές προμήθειας, όσον αφορά τους αγωγούς. Όμως ταυτόχρονα έχουμε όλα αυτά τα έργα, όλες αυτές τις ε, επενδύσεις που πρόκειται να μας κάνουν πολύ πιο εξαρτημένους από την Ρωσία. Είναι πολύ η πολιτική οι οποίες συμφωνούν με τέτοιου είδους σχέδια πολιτικά, εμπορικά και ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα το γερμανικό κράτος είναι κάτοχος, κύριος κάποιων εταιριών οι οποίες προσυπέραψαν τη συμφωνία με την Gazprom. Δεν έλεγε ότι αγνοούσε τις εξελίξεις η γερμανική κυβέρνηση ο South Stream θα εξαφανιστεί. Οπότε και η Βουλγαρία αλλά και η Πολωνία πρόκειται να ε, βλαβούν όπως και η Ουκρανία αλλά και η Τουρκία. Ήδη η Ουκρανία θεωρεί ότι θα έχει ζημία 2 δις ευρώ ετησίως. Και λένε ότι είναι προδοτικό αυτό το πρόγραμμα, ότι προδίδει τα ιδιότητα της αλληλεγγύη. Άρα θα πρέπει να σταματήσει αυτό το έργο, αυτό το έργο κύριε Πρόεδρε. Ο κύριο Γκέρεκ Η Ενεργειακή Ένωση είναι μια ανταγωνιστική αγορά από τη μία, από την άλλη πρέπει και να τηρήσει τους ε, στόχους για το κλίμα. Για να γίνει αυτό πρέπει και να ενισχυθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε και τα δύο. Όταν αν θέλουμε μάλλον να σκεφτούμε λογικά και μακροπρόθεσμα, τότε μπορούμε να δούμε πως υπάρχουν διαφωνίες οι οποίες είναι και ιστορικά αιτιολογημένες. Μπορούμε λοιπόν να κρίνουμε εάν η όχι ότι ο πλασιασμός της χωρητικότητας του North Stream είναι ε, συνετός ή όχι. Ο ενεργειακός εφοδιασμός είναι προτιμότερος να γίνει με, αυτό, ε, με φυσικό αέριο παρά με άνθρακα. Χρειάζεται όμως ε, ευελιξία στην παραγωγή ενέργειας. Γι' αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλες πηγές όπως η αιωλική ενέργεια και να συμπεριληφθούν επίσης και οι ώρες εχμής, για παράδειγμα στην ε, γεωργία. Όλα αυτά είναι γνωστά βέβαια. Κοινά όμως έργα, όπως αυτό, πρέπει να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λαμβάνεται υπόψη και η διαφοροποίηση στα ανατολικά αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της ε, ομάδας ECR έχετε ένα λεπτό καιρό. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο διπλασιασμός της χωρητικότητας του North Stream είναι κάτι που μας βρίσκει αντίθετους. Εμείς θέλουμε να γίνουμε περισσότερο ανεξάρτητοι από το ρωσικό φυσικό αέριο και ταυτόχρονα να ψάξουμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αν δούμε τη χωρητικότητα του North Stream, θα παρατηρήσουμε ότι χρησιμοποιεί μόνο το 50% των δυνατοτήτων του. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να επιτρέψουμε το θέμα αυτό να αναχθεί σε γεωπολιτικό ζήτημα. Το θέμα είναι από πού θέλουμε να λαμβάνουμε την ενέργειά μας στο μέλλον και πού μπορούμε να στηριχθούμε. Χρειάζονται ε, πρώτες ύλες και πρέπει να έχουμε την ε, ασφάλεια αυτών. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν το αέριο για να ασκήσουν επιρροή σε διάφορες χώρες και για να τις σταματήσουν να στραφούν προς την Δύση. Αυτό μας είναι γνωστό. Για παράδειγμα, το 2007 οι αποστολές πετρελαίου προς την Εστονία είχαν ανασταλεί και ταυτόχρονα είχε σταματήσει να πηγαίνει φυσικό αέριο προς την Γεωργία και η Ουκρανία είχε αυξήσει τις τιμές. παρομοίω στην Αρμενία, στην Κυργησία, στην Τρανσνίστρια. Όλα ε, αυτές οι χώρες είχαν επηρεαστεί από την ε, αύξηση αυτή των τιμών, ακόμα και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, Βοσνία, Σερβία κτλ. Θα ήθελα να πω ότι γνωρίζουμε πως ο αγωγός North Stream θα μειώσει την εξαρτήσή μας από την Ουκρανία. Όμως, τι θα γίνει στο μέλλον, την θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθούν τέτοια περιστατικά στο μέλλον. Ο κύριος Λευτέρης Χριστοφόρου έχει το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο οφείλω να τονίσω είναι ότι πρέπει σε αυτή την αίθουσα να είμαι θα όλοι αντικειμενικοί και ειλικρινείς. Τουλάχιστον αυτό το οποίο εγώ ακούω από την ημέρα που εκλέγηκα Ευρωβουλευτής, από όλους, από το Ευρωκοινοβούλιο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον Αρμόδιο Επίτροπο, από τους πάντες είναι ότι οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί ενεργειακά αυτοδύναμη, αυτάρκης, να υπάρξει απεξάρτηση, να υπάρξουν πολλές ενεργειακές πηγές εφοδιασμού, να μην είναι όμοιρος και ελεγχόμενη ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα διασφαλίσουμε. Το αφήνω στην κρίση του καθενός να μας πει αν διασφαλίζεται όλο αυτό μέσα από το Nord Stream 2 αυτό που έχω να πω είναι ότι και σήμερα ο κύριος επίτροπος πολύ ορθά ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να έχει πολλές πηγές εφοδιασμού φυσικού αερίου. πώς επιτυχάνεται όμως αυτό; εδώ είναι η ώρα της κρίσης η ώρα των αποφάσεων και η ώρα των προτάσεων. εμείς έχουμε προτάσεις. μια αξιοποιήσουμε τις εγχώριες πηγές εφοδιασμού. θεωρώ ότι η ανατολική μεσόγειος αλλά και άλλες περιοχές προσφέρονται για την ευρωπαϊκή ένωση να τις αξιοποιήσει και να καταστήσει όσο το δυνατό περισσότερο αυτάρκη και να μην είναι εξαρτώμενη από μία ή από δύο πηγές η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα ενέργειας. Θεωρώ ότι η Ανατολική Μεσόγειος προσφέρεται και μέσω της Κύπρου που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί ένας εναλλακτικός βραχίωνας ενεργειακού εφοδιασμού αξιοποιώντας την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Θεωρώ όμω ότι υπάρχουν και άλλε περιοχέ που μπορούν να δώσουν εναλλακτικέ λύσει και εναλλακτικέ προτάσει εφοδιασμού. Θεωρώ ταυτόχρονα ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε λύσει τέτοιε που δεν θα καταστήσουν για το παρόν και το μέλλον όμοιρο την Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα ενέργεια. Πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε αντικειμενικά με προτάσει που θα έχουν παρόν, μέλλον και προοπτική και μια τέτοια πρόταση είναι επιτέλου να αξιοποιήσουμε την Ανατολική Μεσόγειο προ την ορθή κατεύθυνση και να επενδύσουμε σε ενεργειακέ υποδομέ προ εκείνη την κατεύθυνση προ όφελο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προ όφελο των ευρωπαίων πολιτών προ όφελο του ενεργειακού φοδιασμού και τη αυτάρκεια ενέργεια για την ευρωπαϊκή ένωση. Ευχαριστώ. Έχει το λόγο τώρα ο κύριος Κόφοντ. Κύριε Πίτροπε, κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να επεκταθεί ο North Stream. Τα πράγματα είναι απλά. Η ενεργειακή μας ένωση πρέπει να χτιστεί βασισμένη στην αλληλεγγύη, στη συνεργασία και στην ανανεώσιμη ενέργεια. Και ο North Stream είναι το ακριβώς αντίθετο από όλα αυτά. Ο North Stream δεν περνά από την Πολωνία, παρακάμπτει την Πολωνία, παρακάμπτει τις ευαλτικές χώρες, δεν χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που έχουμε. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε την Ευρώπη και όχι να την αποδυναμώσουμε. Ο Πούτιν που αυτή τη στιγμή βομβαρδίζει τη Συρία δεν αξίζει οποιαδήποτε ανταμοιβή τέτοιου τύπου. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε την εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αντίθετα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ε, ενεργειακή αυτάρκεια και στην δημιουργία μιας σωστής ε, ενιαίας αγοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έργο σας είναι να συμβεί αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιατσκέβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας υπενθυμίσω ότι η χώρα μου, η Πολωνία, από την αρχή των ε, διαβουλεύσεων για τον αγωγό ε, North Stream είχε τοποθετηθεί ξεκάθαρα για τον ε, αγωγό. Το θέμα είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Τα μέτρα όμως αυτά δεν συμφωνούν με τις διατάξεις περί αλληλεγγύης και ενεργειακής αυτάρκειας. Το ευρωπαϊκό δίκαιο αν κοιτάξουμε τις ε, ιδρυτικές ε, αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει το ακριβώς ε, αντίθετο. Αυτό όμως που παρατηρώ είναι ότι οι περισσότεροι σιωπούν για αυτό το θέμα. Η ενεργειακή ασφάλεια και η οικονομία της Ευρώπης είναι αυτά που πρέπει να ενισχυθούν. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι ο αγωγός North Stream το μόνο που θα ενισχύσει είναι το μονοπόλιο της Ρωσίας και θα αποσταθεροποιήσει την ε, ενεργειακή αυτάρκεια ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου του τρίτου ενεργειακού πακέτου. Αυτό είναι κάτι που σας καλώ να αναλογιστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τσάμπα Μόλναρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ κύριε Επίτροπε, δεν είναι σίγουρο το ότι χρειαζόμαστε αποκλειστικά και μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή είναι μια ιδεολογία των πρασίνων. Εδώ μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη, για θέσεις απασχόλησης, για την κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Χρειαζόμαστε και τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας, όμως κυρίως χρειαζόμαστε διαφοροποίηση στην ενέργεια, διότι χωρίς αυτή η ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη δεν είναι βιώσιμη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βλέπουμε ότι οι τιμές της ενέργειας έχουν ε, εξαιτία της διαφοροποίησης και σίγουρα συνεισφέρει το ρωσικό φυσικό αέριο σε αυτό όμως η ενεργειακή μας εξάρτηση δεν θα πρέπει να είναι μονόπλευρη δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εξαρτώμαστε εμείς μόνο από την Ρωσία πρέπει να σκεφτούμε και τι γίνεται από την άλλη πλευρά οι εταίροι μας ε, στην Ανατολή είναι πολύ πιο αξιόπιστοι διότι μας χρειάζονται και χρειαζόμαστε και ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σπίγνιεφ Κούσνοφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το επενδυτικό πρόγραμμα για τον αγωγό North Stream είναι κάτι κυρίως πολιτικό και όχι οικονομικό, διότι αφορά τα πλεονεκτήματα που θα έχει η μία μόνο πλευρά η Μεγάλη Δυτική ομίλη η Gazprom, η οποία θα μπορέσει να επεκτείνει το δίκτυό της. Και παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τίθεται κατά των μονοπωλίων, αυτό που κάνει τώρα είναι μία ένδειξη, μία απόδειξη μάλλον, του ότι καταπατάται η ανεξαρτησία. Οι κυβερνήσεις ε, των κρατών μελών πρέπει να απαιτήσουν αλληλεγγύη από τα άλλα κράτη-μέλη. Και όταν αυτό το κάνουν για το προσφυγικό ζήτημα, τότε παρακαλώ να απαιτήσουν και αλληλεγγύη στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Και όχι μόνο για το συγκεκριμένο έργο, αλλά και ε, να λάβουν υπόψη τις διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσουν αυτές οι μονόπλευρες επενδύσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η ενεργειακή ασφάλεια είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση για την Ευρώπη, διότι στο Ηνωμένο Βασίλειο η εξάρτηση από τι αγωγέ έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδίω δε όσον αφορά το φυσικό αέριο. Και στα πλαίσια αυτά θα ήθελα εγώ να σα τονίσω ότι η λύση όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια είναι και το να δούμε πώ θα εμφαθύνουμε την ολοκλήρωση τη αγορά πώς θα ισχυροποιήσουμε τις προσπαθίες μας, θα τις εντείνουμε σε την αποτελεσματικότητα και πώς θα έχουμε την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το να διπλασιαστεί η παροχή από αυτόν τον αγωγό σημαίνει διάφορα πράγματα τα οποία θα πρέπει προσεκτικά να αξιολογηθούν. Πρώτα-πρώτα, κύριε Κανιέτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει το ότι αυτό το έργο συνάδει προ τα όσα ισχύουν στο, ενεργικό, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τι Ενεργειακέ Αγορέ. Παρακαλώ την Επιτροπή να ερευνήσει ταχύω αυτή διπλασιασμό τη παροχή, τι πάει να πει για για ε, τις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Διότι είναι προς το συμφέρον μας να μπορούμε να βρούμε μια ε, συνολική λύση για την ενεργική ασφάλεια και έτσι να μπορέσουν να ωφεληθούν όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ δεν έχω πιστεί ότι αυτό το έργο είναι μέρος μιας λύσης. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα, προχωρούμε στην διαδικασία Catch the Eye, ελκύω την προσοχή του Πρόεδρου. Έχουμε εδώ ένα πολύ μακρύ κατάλογο. Ο κύριος Χέντμαν πρώτα θα λάβει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε όλα απόψε. Οπότε και εγώ ας περιοριστώ εις το πιο σημαντικό, εις την αλληλεγγύη και τον σεβασμό, την τήρηση του δικαίου. Αυτά είναι το θεμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πρόσφατα έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το σημερινό θέμα και απόψε επίσης χίλιες φορές αναφέραμε αυτές τις αρχές μα η αλληλεγγύη δεν θα πρέπει να είναι κάτι δεσμευτικό για όλους και από την άλλη μεριά είναι δυνατόν να έχουμε ένα τέτοιο ζήτημα σαν το Nord Stream το οποίο να το απορρίπτει κανείς σε σχέση με την οικονομική του ε, αποτελεσματικότητα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την αντίθεση. Σας ευχαριστούμε κύριε Βουλευτά, λέει ο Πρόεδρος. Φραντζούλητσα. Κύριε Επίτροπε, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2014 θεώρησε ότι θα πρέπει να καταρτήσουμε ένα σχέδιο για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία, πέρα από τη χρήση άλλων προμηθευτών εκτός Ρωσίας, ένα στόχος θα πρέπει να είναι να χρησιμοποιήσουμε νέες ενεργειακές πηγές. Ο φυσικός αγωγός North Stream θα έπλητε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Θα τασόταν υπέρ ορισμένων ευρωπαϊκών πολιεθνικών και θα μείωνε την αλληλεγγύη που η Επιτροπή πρόβαλε μετά από σύσταση των κρατών μελών. Επίσης, πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα τάσσονταν κατά της αλληλεγγύης και της συνοχής. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να σταθούμε στην ενεργειακή στρατηγική ασφαλείας έτσι ώστε να μην υπάρχουν εμπορικές διαφορές και να μην καταρρύψουμε τις υποδομές που ήδη υπάρχουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο nord stream 2 αποδεικνύει ότι και στον ενεργειακό τομέα η οικονομία καθορίζει τις αποφάσεις. την ίδια ώρα που η κυρία μέρκελ διαβεβαίωνε ότι δεν θα εγκαταλείψει την ουκρανία οι γερμανικές εταιρείες μαζί με άλλες ευρωπαϊκές πολυεθνικές έκλειναν με την gazprom τη συμφωνία για τον διπλασιασμό του δυναμικού του nord stream. το πράττουν αυτό διότι θεωρούν ότι είναι η φθηνότερη λύση. οι επιχειρήσεις αλλά και κυρίως οι καταναλωτές έχουν ανάγκη από πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να διαφοροποιηθούν τόσο οι πάροχοι όσο και κυρίως οι ενεργειακοί δρόμοι. η στρατηγική των πολλαπλών νότιων ενεργειακών διαδρόμων και το πέρασμά τους από την πατρίδα μου την ελλάδα είναι κομβική σημασία σε αυτό το θέμα. με τις εξελίξεις στο ιράν την κατασκευή του ΤΑΠ, την ανακάλυψη των κοιτασμάτων σε αίγυπτο ισραήλ κύπρο και με τα κοιτάσματα στην ελλάδα το ενεργειακό πλαίσιο αλλάζει άρδιν η ελλάδα πρέπει να αποτελέσει στρατηγικό ενεργειακό κόμβο και πύλη εισόδου στη νέα αρχιτεκτονική αξιοποιώντα τα ενεργειακά αποθέματά της μακριά από την κυδαιμονία της τρόικα και των δανειστών με μόνο γνώμονα το όφελος του λαού μας και την ευημερία του. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να βλέπει την υπόθεση αυτή μόνο σαν κομμάτι της εμπορικής πολιτικής. Θα πρέπει να δίνεται το ευρύτερο τοπίο, την αλλαγή του κλίματος, την ενεργειακή πολιτική και τους στόχους της. Γιατί είναι προφανές ότι αντιβαίνει στους σκοπούς μας. Δεν ωφελεί όσον αφορά το να έχουμε ποικιλία στην προμήθεια της ενέργειας αυτό το έργο δεν, δεν, δεν συνάδει και προς τις προτεραιότητές μας. Θα πρέπει επομένω να δούμε τι θα κάνουμε για να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια. Υποδομές στην ε, ε, Βαλτική μα έχουμε εναλλακτικέ όσον αφορά την ε, πρόμηθη ενέργεια. Α, στη Λιθουανία έχουμε ένα τερματικό υγροποιημένο φυσικό αέριο και ελπίζω ότι το έργο αυτό τελικά δεν πρόκειται να οδηγήσει σε ένα καινούριο βατερλό της πολιτικής μας. Δεν θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον της ενεργικής πολιτικής μας. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξουμε τέτοια σχέδια και προγράμματα. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ο Επίτροπος. Μιγέλ Άριας Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι βουλευτές, να σας ευχαριστήσω όλους για τις παρατηρήσεις σας. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Στα πλαίσια της ειδικής ασφάλειας, ναι, χρειάζεται να υπάρχει διαφοροποίηση. Να, ποια είναι η πολιτική την οποία εμείς έχουμε χαράξει. Είμαστε υπέρ όλων των σχεδίων που συνάδουν προς αυτή την πολιτική στρατηγική και για το φυσικό αέριο. Αυτό ξεκίνησε φέτος και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το εγκροπημένο φυσικό αέριο έτσι να ε, το χειριστούμε στο μέλλον. Και είμαστε υπέρ αυτών των εξελίξεων ε, εις τον νότιο διάδρομο. Ο τουρκικός αγωγός ε, θα έχουμε 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα περάσει από το Αζερμπατζάν το Τουρκμενιστάν και θα έχουμε κάποια στιγμή και φυσικό αέριο από το Ιράν. Έχουμε εξελίξει τώρα στην Μεσόγειο. Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Περίπου 3.000 BCM που έχουν ε, βρεθεί σε κοιτάσματα και υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που διαφαίνονται. Θα πρέπει επίση να δούμε πώς ε, θα ε, έχουμε ε, παροχή και προς την κεντρική Ευρώπη. Άρα υπάρχει τώρα ε, αυτή η πολιτική της, ε, της διαφοροποίησης. Οπότε και αυτός ο δεύτερος αγωγός Nord Stream συνάδει, δεν έρχεται σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική. να τον φτιάξουμε δεν θα έχουμε εξάρτηση από έναν προμηθευτή και θα έχουμε και περισσότερες οδούς γιατί βλέπουμε ότι θα περάσει από την Ουκρανία και θα έχουμε 80% των εισαγών του ρωσικού αερίου. Από μία διαδρομή θα έχουμε κυρίαρχη θέση της Gazprom στη γερμανική αγορά και από το 40% θα πάει στο 60% το κομμάτι της αγοράς. Οπότε το να ευθυγραμμιστεί αυτό το έργο με την στρατηγική μας για την ασφάλεια ε, γεννεί κάποιες εμβολίες. Οπότε και για αυτό θα πρέπει να έχουμε ασφαλή διέλευση από την Ουκρανία όπου τώρα έχουμε το φυσικό αέριο που έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε υπερβολική παροχή από την Ρωσία τώρα. Οπότε και γι' αυτό το Nord Stream 2 δεν μπορεί να είναι κάτι κοινού ενδιαφέροντος και δεν μπορεί να ωφελήσει ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε την προσεκτική αξιολόγηση αυτού του έργου του Nord Stream 2 και θα λάβουμε υπόψη ό,τι ισχύει σήμερα. Να δούμε τι γίνεται με τη ρυθμιστική αρχή της Γερμανίας. Να δούμε στις λεπτομέρειες αυτό το έργο. Οπότε και γι' αυτό θα εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την νομιμότητα αυτού του έργου και πρόκειται να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε εξελίξεις. Θα πρέπει οι εταιρείε να αποφασίσουν αν είναι βιώσιμο αυτό το έργο ή όχι. Αλλά ε, θα πρέπει να δούμε το πώς το θα, θα τηρηθεί το κοινωτικό κεκτημένο. Όπως είπα πριν, το Nord Stream 2 θα πρέπει να συνάδει προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά το τρίτο πακέτο για την ενέργεια του σιδηρόδρομου. Επίσης, εγώ θα ε, φροντίσω προσωπικά να ισχύσει αυτό που σας λέω. Ο Πρόεδρος. European Council. Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κύριος Νικολά Σμιτ, ε, εντάχει κύριε Πρόεδρε. Η Προεδρία ευχαριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την τόσο χρήσιμη συζήτηση και για τη σημασία που προσδίδει στο θέμα του ενεργειακού εξοπλισμού και ασφάλειας. Η ενεργειακή ασφάλεια και ανεφοδιασμός είναι ύψης της σημασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η ενεργειακή ασφάλεια, όπως έδειξε και η συζήτηση, ενέχει πολλά στοιχεία οικονομικά, περιβαλλοντικά αλλά και γεωπολιτικά. Θα πρέπει να προωθήσουμε κοινούς στόχους και να μιλήσουμε με μία φωνή. Η Ευρώπη της ενέργειας θα δώσει μία πλαισίωση ε, έργου και εργασίας για να φτάσουμε στους στόχους μας. Με βάση αυτά που είπε ο Επίτροπος, θα ήθελα να σας αναφέρω τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ης Μαρτίου 2015. Το σημείο Δέλτα που αναφέρει θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε η αγορά φυσικού αερίου να συμβαδίζει με το κοινοτικό δίκαιο, ιδιαίτερα ενισχύοντας τη διαφάνεια αυτών των συμφωνιών και τη συμβατότητά τους με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτά που μας προείπε ο Επίτροπος κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό θα διαβιβάσουμε τις ανησυχίες που αναφέρατε σε εκείνους που πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ τον